We start the meeting with adoption of the agenda. Αρχίζουμε τη συνεδρίαση με, την ε, έγκριση της σημερινής διάταξης, η οποία θα εγκριθεί με τις εξής ε, αλλαγές. Έχουμε στο σημείο υπαριθμών 8 που έχουμε αυτή τη σύσταση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για, για ε, το TTIP θα γίνει πριν το 4. Πριν το 4, το οποίο είναι η πρόταση οδηγίας Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με τους ναυτικούς που τροποποιεί μια σειρά οδηγιών. Τώρα, το σημείο υπαριθμών 2, ανακοινώσει τη Προέδρου. Κλείνει το μικρόφωνο. Όχι, εκτός μικροφώνου μιλάει κάποιος. Do the interpretation works now? Α, λειτουργούν τα μικρόφωνα τώρα ε, ε, για να ακούμε τη διερμηνία. Καλώς. German too, uh, Is there a technical problem with the... Υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα, δεν ακούτε κάτι. Με την γερμανική ε, καμπίνα υπάρχει ένα πρόβλημα, το μικρόφωνο τους σβήνει, λέει η κυρία βουλευτής. Do we know if the, the German... Now it works. Now Τώρα, α, εντάξει λέει η κυρία Στάινμπρουκ, τώρα λειτουργεί, ακούγεται η γερμανική καμπίνα. Ε, για τώρα, ανακοινώσει πρόεδρου, θέμα υπαρθμών 2. Τι, θα σα πω ότι έχουμε όλε τι γλώσσε εκτό από φιλανδικά, κροατικά και μαλτέζικα. Και κατά δεύτερο λόγο, σα ενημερώνω ότι η γραμματεία από 2 Απριλίου μέχρι 12 Απριλίου ε, έχει ε, έργα στα οποία περνάει ο χώρος οπότε θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι το σχετικό προσωπικό ή το σχετικό και οι συνεργάτες έχουν μετακινηθεί σε κάποιους άλλους χώρους για λίγο. Πάμε τώρα στο θέμα υπαριθμών 3 της σημερινής διατάξεως το οποίο αφορά τις μονοπρόσωπες εταιρείε περιορισμένης ευθύνης. Και θα δώσουμε το λόγο τώρα στην εισηγήτρια, την κυρία Γιούτα Στάινμπρουκ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Προτείνω στην Επιτροπή Απασχολήσεως να παραπέμψει, να ζητήσει την απόσυρση δηλαδή της οδηγίας διότι πρόκειται για, νέο, για επανάληψη του σχεδίου της Ευρωπαϊκής Εταιρεία που είχε επικριθεί τότε από το Κοινοβουλίο και αποσύρθηκε τελικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εξακολουθούν να υπάρχουν τα ίδια προβλήματα. Προωθείται η δημιουργία με, τον, με την πρόταση αυτή των περίφημων εταιριών γραμματοκιβωτίου και καταρχήν βέβαια η η ιδέα είναι καλή, να διευκολυνθεί δηλαδή η ίδρυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αλλά δεν επιτυγχάνει το στόχο της. Δεν περιορίζει το πεδίο εφαρμογής σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν προϋποθέτει ότι θα πρόκειται για διαμεθοριακή συνεργασία για την ίδρυση επιχειρήσεως. Υπάρχει και διάκριση μεταξύ, χωρισμός δηλαδή μεταξύ ε, έδρας και καταστατικού. Δεύτερο, ε, καταχώρηση στην ε, επιγραμμικά και ούτω καθεξής. Και πάνε να φτιάξουν δηλαδή ένα δούριο νύπο που δεν οδηγεί σε βιώσιμες δραστηριότητες μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στην ουσία κάνουν δώρα σε επιχειρήσεις που αποκομίζουν κέρδη μόνο δια της φόρο αποφυγής με ναι, εταιρείε γραμματοκιβωτίου. Και σε αυτή την κρίση συμφωνούν πολλοί και από τους ενδιαφερομένους στα δίκτυα αυτά και συνδικάτα και ενός εργοδοτών και συμβουλόγραφοι αλλά και ίδια η Ένωση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Τώρα έχω τρία σύντομα σχόλια που παίζουν σημαντικό ρόλο για να ζητήσω την απόρριψη. Πρώτα λοιπόν για τη χώρα καταχώρησης της SUP ανεξαρτήτως του που δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Αυτό σημαίνει ότι καταστατηγούνται οι διατάξεις προστασίας ορισμένων χωρών μελών, ορισμένων νόμων τάξεων με τον τρόπο αυτό ανοίγονται παράθυρα για φοροαποφυγή με ψεύδο αυτοαπασχόληση και αυτό οδηγεί σε ζημιά και των φορολογικών εισόδων των χωρών μερών και των κοινωνικών συστημάτων. Δεύτερο, το ελάχιστο κεφάλαιο. Η πρόταση δεν προβλέπει ελάχιστο κεφάλαιο, ούτε δημιουργία αποθεματικών. Και επομένως δεν υπάρχει η απαραίτητη χρηματοδοτική βάση για εταιρείε με περιορισμένη ευθύνη, που είναι απαραίτητη για τις συναλλαγές. Πρόκειται εν τέλει για την προστασία των δανειστών τους, αλλά και των απαιτήσεων των εργαζομένων. Τρίτο είναι η επιγραμμική, online δηλαδή, καταχώρηση. Υποτίθεται ότι θα οδηγήσει ως σε ελάφρυνση της γραφειοκρατίας. Όμως ανοίγει το δρόμο για διάφορες παράνομες δραστηριότητες. Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, ε, απατηλή πτώχευση και ούτε καθεξής. Ώστε να μην υπάρχει χρήμα για να ικανοποιηθούν εκ των υστέρων οι Ο χαρακτηρισμός SUP υποτίθεται ότι θα είναι παντού ο ίδιος, αλλά αυτό δεν εξασφαλίζει ασφάλεια δικαίου. Αυτά ως συγκρότηση για την απόρριψη. Ε, thank you. Ε, Σας ευχαριστώ λέει Πρόεδρος. Και τώρα να ακούσουμε τους πιο δεσηγητές. Κύριος Μπέκερ, από το ΕΛΚ. Κύριε Μπέκερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν επιθυμώ και εγώ να εκφράσω την συμφωνία για αυτήν την πρωτοβουλία. Έχει νόημα όντως να προσανατολιστούμε προς τα εκεί. Νομίζω η ίδρυση επιχειρήσεων αποτελεί μέρος των μελλοντικών οικονομικών εξελίξεων, δηλαδή που θα επηρεάσει θετικά τις μελλοντικές οικονομικές εξελίξεις. Επίσης πιστεύω ότι τα βασικά δεδομένα, ελάχιστο κεφάλαιο, προστασία εργαζόμενων κλπ. δεν ρυθμίζονται ικανοποιητικά στην πρόταση. Νομίζω ακόμη ότι δεν έχω βέβαια τόσες πολλές αντιρρήσεις ιδεολογικο-αριστερές όπως η συναδελφός μου που προλάβησε, αλλά θα συμφωνήσω με την πρότασή της, διότι μπορούμε να περιμένουμε, είναι πιο λογικό τι θα πει η νομική επιτροπή, νομίζω είναι πιο λογική αυτή η διαδικασία, διότι εκεί νομίζω οι βουλευτές δουλεύουν σε βάθος, με σοβαρότητα, εξετάζουν όλα τα θέματα και του ελάχιστου κεφαλαίου δηλαδή κτλ. ώστε είναι σωστό νομίζω, κατά εξαίρεση, να περιμένουμε για μια φορά ω Επιτροπή Απασχολήσεω το τι θα πει κάποια άλλη κοινοβουλευτική επιτροπή και μετά να εξαγάγουμε τα συμπεράσματά μα ή να τα συναγάγουμε. Δεν έχει μικρόφωνο η πρόεδρο. Ευχαριστώ κύριε Κράσινοντεύσκη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να σας πω ότι συμφωνώ με κάποιες από τις ε, επιφυλάξεις της εισηγήτριας. Εδώ λείπουν κάποιες ασφαλιστικές δικλίδες όσον αφορά τις ε, εταιρείε ε, γραμματοκιβώτιο και όσον αφορά το ελάχιστο κεφάλαιο. Άρα θα πρέπει να το σκεφτούμε καλύτερα και πολλές φορές τα έχουμε συζητήσει. Θα πρέπει να σκεφτούμε το ότι η Ευρώπη διαφέρει πολύ από χώρα σε χώρα αφορά τις ρυθμίσεις για αυτά τα ζητήματα. Ας πούμε τις ε, ε, εισφορές. Είναι διαφορετικά ρυθμισμένο αυτό σε κάθε χώρα. Επίσης και το κοινωνικό dumping πολλές φορές συντρέχει. Μα η οικονομική πραγματικότητα σε κάθε χώρα είναι τελείως διαφορετική. Άρα θα πρέπει να κάτσουμε και να σταθμίσουμε. Από τη μία μεριά πώς θα έχουμε πιο εύστοχη νομοθεσία και από την άλλη μεριά θα πρέπει να εξασφαλίσουμε το ότι αυτή η πρόταση να είναι τέτοια που να βοηθά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε κεντρική και αντολική που έχουν τόσο σημαντικές για την οικονομία. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος η φιλελεύθερη Ο κύριος Γκούκα. Ή μήπως κάποιος άλλος εκπροσωπεί την άλλη. Καλώς. Τότε πάμε ε, στην Γκουε. Κάρι. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την εισηγήτρια. Εξαιρετικό το σχέδιο κειμένου. Συμφωνώ με όλα όσα είπατε και την απογοήτευσή σας με τις επιφυλάξεις σας σε σχέση με το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να διευκολύνει την ίσπραξη των φόρων, δεν θα έπρεπε να δυναμητίζονται τα κοινωνικά δικαιώματα, των εργαζομένων. Συμφωνώ. Θα πρέπει να απορριφθεί η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συμφωνώ με την γνωμοδότηση. Ε, thank you. Our Greens represented by uh, Madam Reinke. Και η πράσινη τώρα. Λείπει η πραγματική μας χειώδηση συγχυτρία. Συμφωνούμε πάντως, είναι γεγονός αυτό, με πολλά από τα όσα λέχθηκαν ως ομάδα των πράσινων. Θεωρούμε και εμείς ότι η πρόταση δεν τηρεί τα υπεσχημένα να δημιουργήσει δηλαδή ένα λαμπρό μέλλον για τις μικρές και μεσέ επιχειρήσεις. Αντίθετα θεωρούμε ότι κρύβει πολλούς κινδύνους. Ορισμένοι εξήγησαν ήδη για ποιους λόγους. Γίνεται πιο εύκολο να ιδρυθούν ψεύτικες εταιρείε που είναι απλά ένα γραμματοκιβώτιο και που αποφεύγουν τους ελέγχους. Δεν επιτυγχάνεται η ανεξαρτησία. Μπορεί έτσι να υπονομευθεί η συναπόφαση των εργαζόμενων. Όλα αυτά οδηγούν να πιστεύουμε ότι χρειάζονται σημαντικότατες βελτιώσεις. Ασφαλώς, καταρχήν είμαστε θετικές απέναντι στην υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, δεν χωρεί αμφιβολία, αλλά δεν υποστηρίζει η πρόταση αποκλειστικά μικρές και μεσές επιχειρήσεις και νομίζουμε ότι ειδικά σε θέματα απόσπασης εργαζομένων, ούτως ή άλλως τα τελευταία χρόνια έχουμε καταβάλει αγώνα για να πληρώνονται τελικά οι εργαζόμενοι, να μην υπονομεύονται τα κοινωνικά τους δικαιώματα με ίδρυση εταιριών γραμματοβικιωτίου, ψεύτικων δηλαδή εταιριών και με άλλους τρόπους. Νομίζουμε ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ουσία ανατρέπει τα αποτελέσματα αυτού του αγώνα. Γι' αυτό συμφωνούμε με τις ε, βουλευτέ που μίλησαν προηγουμένω και ζητούμε και εμεί απόρριψη τη πρόταση τη Επιτροπή. Ο κ. Μπροκ. Συμφωνώ με τον Πολωνό συνάδελφο που είπε ότι όντω πρέπει να δοθούν περισσότερες ευκαιρίες για την ίδρυση μικρών και μεσών επιχειρήσεων. Όμως δεν είναι ξεκάθαρα για μένα τα πλονεκτήματα που υποτίθεται προκύπτουν από το την εδώ την ρύθμιση, έτσι ώστε να ξεχάσω ποια είναι τα αρνητικά. Στην Ευρωπαϊκή Ενιαία Αγορά κάθε επιχείρηση, κάθε μορφής θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιεί την Ενιαία Αγορά. Δεν μου έχουν εξηγήσει λοιπόν τι προσφέρει αυτή η ε, νέα πρόταση. Υπάρχουν ωστόσο, ελοχεύουν οι κίνδυνοι που επεσήμαναν οι διάφοροι συνάδελφοι. Εταιρείε ψεύτικες με υπονόμευση των δικαιών των εργαζομένων. Αυτά για μένα είναι ε, σαφές ότι εμπεριέχονται. Δημιουργώντα μια τέτοια εταιρεία υπάρχει ο κίνδυνος να υπονομευθούν εθνικά ρυθμισμένα δικαιώματα εργαζόμενων. Εάν τελικά ε, τον τρόπο αυτό τον, τα δικαιώματα των εργαζόμενων, τότε την έχουμε πατήσει. Αυτό λοιπόν ε, με οδηγεί στο να υποστηρίξω την πρόταση της εισηγήτριας να ξαναστείλουμε όλο τον φάκελο στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή να του ζητήσουμε να ξαναμελετήσουν το θέμα, να επανέλθουν γιατί δεν είναι τρόπος αυτός. Ο κύριος Μαν. Βρήκα το κουμπί του μικροφόνου, κυρία Πρόεδρε, μην ανησυχείτε. Ο κύριος Μπέκερ έχει δίκιο. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε ίδρυση επιχειρήσεων. Όχι βέβαια με κάθε τίμημα. Είναι σαν να πούμε ότι θέλουμε πολλές θέσεις απασχόλησης. Θέλουμε βέβαια πολλές θέσεις απασχόλησης, αλλά ποιοτικέ και όχι αβέβαιες. Εάν πάμε να φτιάξουμε επιχειρήσεις με οποιοδήποτε τίμημα, τότε φτάνουμε σε οργανώσεις one man ή one woman και τίποτα άλλο. Εάν δεν διατυπώνεται καν απέτηση για ελάχιστη κεφαλαιοποίηση. Εάν μπορεί κανείς απλούστατα έτσι να καταχωρίζει μια επιχείρηση επιγραμμικά online δηλαδή, στο διαδίκτυο. Αυτό σημαίνει αποφυγή ανάληψης ευθυνών και μπορούν, έχει δίκιο εκεί ο συνάδελφος Πούχατ, ότι δεν προχωρούμε. Παλέψαμε πολύ για την οδηγία απόσπασης εργαζόμενων. Έμα και δάκρυα χύσαμε. Πολλά πετύχαμε υπέρ των εργατριών και εργατών. Δεν μπορούν αυτά τώρα να ανατραπούν. Έχουμε ένα σύστημα κοινωνική οικονομία της αγοράς. Αυτό το κοινωνικό εδώ δεν το βλέπω καθόλου. Το να φτιάχνουν μαζικά επιχειρήσεις αυτό δεν μου αρέσει. Θέλω να κάνουμε ένα επικοδομητικό διάλογο με τους ε, συναδέλφους της Επιτροπής Νομικών. Δεν είναι όλοι αποστεγνωμένοι δικηγόροι που το μόνο που σκέφτονται είναι οι παράγραφοι και οι τελείες και τα κόμματα. Ίσως με κοινή προσπάθεια να καταλήξουμε σε κάποια λογικά αποτελέσματα. Έχω δει αυτά τα πράγματα μιλώντας και με προσώπους εργαζόμενων αλλά και μικρών και μεσών επιχειρήσεων και όλοι μου είπαν διώχτε το αυτό το, διώχτε την πρόταση ευχαριστώ Thank you, Madam President. Να πω και εγώ με τη σειρά μου ότι είμαι πάρα πολύ απογοητευμένος ε, από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διότι όταν κάναμε την ακρόαση για τους ε, επιτρόπους έθεσα στον κύριο Ντομπρόσκι μία ερώτηση ακριβώς για αυτό το ζήτημα. Τον ρώτησα για τους κινδύνους της μονοπρόσωπης εταιρεία σε σχέση με τα εργασιακά δικαιώματα και άλλες αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει αυτή η μορφή επιχείρησης. Δεν έκανε τα μαθήματά του, από ό,τι φαίνεται. Δεν είχε κάνει μόνο τα μαθήματά του, γιατί ξαφνιάστηκε από την ερώτησή μου. Μου είπε όμως ότι θα μελετήσει το ζήτημα και με διαβεβαίωσε ότι θα μου απαντήσει με, ε, τον με κατάλληλο τρόπο. Ε, ο κύριος ε, Μπροκ το ζητάει από τον κύριο Ντομπρόφσκι να πάει να κάνει τα μαθήματά του. Ο κύριος Μάν μας μιλάει για την, την κοινωνική οικονομία και από ό,τι φαίνεται το πρόβλημα είναι πολύ βαθύτερο από ότι απλώς μια ενημέρωση του κυρίου Ντομπρόφσκι για το ζήτημα αυτό. Ευχαριστώ. Θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα τώρα, γιατί μετά θα αρχίσουμε τις ψηφοφορίες. Α, η κυρία Στάνιμα. Yeah, Ευχαριστώ τις και τους συναδέλφους για την ευρεία υποστήριξη που χορήγησαν στις ιδέες μου. Πράγματι βρίσκομαι σε στενή επαφή με τις συναδέλφους και τους συναδέλφους της Νομικής Επιτροπής που εξετάζουν και την κοινωνική διάσταση, τι επιπτώσεις της χώρες μέλη, αλλά και στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Και επιπτώσεις θα υπάρξουν βεβαίως ε, σε βάρος των εργαζομένων. Αυτά δεν έχουν σχέση με αριστερές ιδεολογίες, κύριε Μπέκερ. Η επιθυμία απόρριψης της προτάσεως προέρχεται κυρίως από τι ενώσεις μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Δεν περιορίζεται άλλωστε η πρόταση της Επιτροπής σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και μεγάλοι όμιλοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη ρύθμιση αυτή, είτε νομίμως είτε και παρανόμως, αλλά και νομίμως. Δεν περιορίζεται βεβαίως η νομοθετική αυτή ρύθμιση στις μικρές επιχειρήσεις, ούτε πρόκειται μόνο για ίδρυση μικρών μεσαίων επιχειρήσεων και διορτάται κανεί, αν όντω θα δημιουργηθούν έτσι θέσει απασχολήσεω ή τέλο πάντων με ποιο, τρο... με ποιο σκοπό θα ιδρύονται SUP. Ευχαριστώ πάντως για τη συζήτηση που διεξήχθη. Θα διατηρήσω επαφή και με τους σκιώδει συγητέ και οι εισηγητρίες καθώ και με του συναδέλφου τη Νομική Επιτροπή, ώστε να καταλήξουμε σε ξεκάθαρε θέσει. Όμω, συμβάλλουμε και στο έργο της Νομικής Επιτροπής εάν τους δώσουμε και εμείς ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Σας ευχαριστώ. Έχουμε και χρόνο να ακούσουμε τον κύριο Κόρτς από τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Just, αν θέλετε. Ευχαριστώ. Ε, είναι μάλλον απογοητευμένα τα μέλη της Επιτροπής και εμείς το ίδιο διότι ε, στην ΙΜΚΟ και στη Γιούρη είχαμε την ευκαιρία τουλάχιστον να παρουσιάσουμε την πρότασή μας. Αν είχα, μας είχε δοθεί αυτή η ευκαιρία θα είχαμε ίσως ε, διευκρινίσει κάποιες παρανοήσεις που έχουν προκύψει μεταξύ των οποίων και ζητήματα που έθεσε η συγγήτρια. Με έκπληξη ακούσαμε ότι υπάρχουν ανησυχίες που δεν αιτιολογούνται ε, από το περιεχόμενο της πρότασης σε σχέση, παραδείγματος χάρη με την επιγραμμική εγγραφή. Είναι ξεκάθαρο στην πρότασή μας ότι το κράτος μέλος όπου γίνεται η εγγραφή ελέγχει την εγγραφή. Δεν τίθεται ζήτημα να δημιουργηθούν ε, εικονικές επιχειρήσεις υπάρχουν ασφαλείς διαδικασίες ε, επιγραμμικής εγγραφής ε, που λειτουργούν ε, εύρυθμα σε 16 κράτη-μέλη. Το θέμα της φορολογίας είναι ξεχωριστό. Δεν σχετίζεται άμεσα με το αντικείμενο της πρότασης. Η νομολογία του δικαστηρίου εδώ και χρόνια επιτρέπει το διαχωρισμό των δύο χωρών, δηλαδή της έδρας και του καταστατικού ε, και ε, σε χώρες όπως αυτή της εισηγήτριας επιτρέπεται ο διαχωρισμός αυτός ε, και ο διαχωρισμός αυτός κατά αυτός δεν δημιουργεί φορολογικά προβλήματα. η χώρα της κυρίας έδρας ε, είναι ε, και ε, η χώρα όπου είναι η η εταιρεία και κυρίως εκεί πέρα που καταγράφονται τα κέρδη της επιχείρησης. Ήθελα να εξηγήσω και άλλα τέτοια στοιχεία της πρότασης, αλλά πολύ φοβάμαι ότι δεν έχω χρόνο τώρα να το κάνω, οπότε θα σταματήσω. Κυρία Ουλσκόγκ, ευχαριστούμε κυρία Στάινλουκ για το επιχείρημα ότι ο διαχωρισμός έδρας υπάρχει ίδιος ρύθμιση σε πολλές χώρες μέλη και η παραπομπή στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Ναι, στην απόφαση του το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αναγνωρίζει καταρχήν την εγκατάσταση σε άλλη χώρα. Όμως την περιορίζει σε πρόσφατη απόφασή του σημαντικά, διότι τώρα το ΔΕΚ ζητεί ότι η δραστηριοποίηση σε, στην χώρα της καταχώρησης έχει ως στόχο να περιορίσει και ε, προσπάθειες φοροαποφυγής κτλ. Αυτό κατέστησε σαφές και στις συζητήσεις που διεξήγαγα εγώ. Δηλαδή και εκεί το ΔΕΚ έχει προβεί σε βελτίωση της ομολογίας του. μπορώ να παραπέμψω και σε πολλές συζητήσεις, μελέτες και αναλύσεις και των επιπτώσεων και σε πολλές χώρες μέλη. Thank you. We will now... Ευχαριστώ. Θα προετοιμαστούμε τώρα για τις ψηφοφορίες. Ah, okay, I have to repeat the timetable for uh, the, this report. Deadline for amendment. Τώρα για τις μονοπρόσωπες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ε, η Τετάρτη Μαΐου 12 το μεσημέρι είναι η προθεσμία για τις τροπολογίες. Στις 28 Μαΐου θα ε, τις εξετάσουμε. Στην ε, Επιτροπή Απασχόλησης στις 23 Ιουνίου θα ψηφίσουμε για την έκθεση και στη Γιούρη στις 15 Σεπτεμβρίου, το φθινόπωρο. Ας προετοιμαστούμε τώρα για τις ε, ψηφοφορίες, γιατί έχουμε πάρα πολλές εκθέσεις να ψηφίσουμε. Ah S'il vous Κυρία Πρόεδρε, πριν αρχίσουμε να ψηφίζουμε, παρακαλώ μια παρατήρηση. Είμαι νέος ευρωβουλευτής μεν και ίσως θα χρειαστεί να συνηθίσω πρώτα, αλλά δεν μπορώ να δεχτώ η λίστα ψηφοφορίας να μην μας διαβιβάζεται ούτε καν 24 ώρες πριν. Χτες το βράδυ στις 10 και 21 λεπτά έλαβα την λίστα ψηφοφοριών. Ε, δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή, πραγματικά δεν είναι δυνατόν. Θα πρέπει πραγματικά να σκεφτούμε ξανά αν μπορούμε έτσι να εργαστούμε. Διότι τα πράγματα που καλούμαστε να ψηφίσουμε σήμερα δεν είναι και ασήμαντα. Κύριε Μαρτά, ευχαριστώ Πρόεδρε. Την ίδια παρατήρηση θέλω να κάνω κι εγώ. Και όχι μόνο αυτό, για το σημείο 8 δεν έχουμε πάρει καν κατάλογο ψηφοφορία. Αν μπορεί η γραμματεία να μας το δώσει ή να μας πει τουλάχιστον τι έχει συμβεί. To Mr. Uh, it was sent to... Uh, Κύριε Μαρτά, να σας απαντήσω. σας το στείλαμε. Η Αναστασία Μητρονάτσιου πήρε εχθές τον κατάλογο στο ηλεκτρονικό της ε, ταχυδρομείο, οπότε κανονικά έπρεπε να το έχετε λάβει. Για τους υπολείπους που αναρωτήθηκαν γιατί αργήσαμε τόσο πολύ, θα απαντήσω ότι συνεχίζονταν συζητήσεις πολιτικές ομάδες για να καταλήξουμε σε συμβαστικές λύσεις. Έτσι έχει πολιτικός βίος στο Κοινοβούλιο, ορισμένες φορές ε, έχει ως αποτέλεσμα να είναι πολύ στενά τα χρονικά περιθώρια. Τα καταφέραμε όμως, Και έχουμε τον κατάλογο και έχουμε και χρόνο στη Κύριε Μάν. Ο κύριος Τόμας Μάν. Νομίζω ότι πρέπει να λάβουμε, οφείλουμε να λάβουμε σοβαρά υπόψη τις επιφυλάξεις των συναδέλφων. Ε, έκθεση της κυρίας Χάρκιν για την συμφωνία TTIP. Εκατοντάδες, να μην πω χιλιάδες, email έχουμε λάβει. Εάν πάμε τώρα σαν τρελή να τα περάσουμε. Οι σκιώδεις ηγητές μας έχουν προσπαθήσει να καταλήξουν σε συμβιβασμούς, δεν το κατάφεραν σε όλες τις περιπτώσεις. Αν δεν είμαστε εις θέση να ελέγχουμε το τι ψηφίζουμε, δεν είναι αποτελεσματική η εργασία μας. Τουλάχιστον δεν είναι δυνατόν αυτή η ψηφοφορία για την έκθεση Χάρκιν να αναβληθεί για την επόμενη ε, συνεδρίαση. Δεν υπάρχει τέλος πάντων και τόσο μεγάλη βία θέλω να γνωρίζω σε κάθε τμήμα πώς έχουν καταλήξει σε συμβαστικέ τροπολογίες. Είναι δυνατόν να αναπληθεί αυτή η ψηφοφορία. Δεν μας επιτρέπει το χρονοδιάγραμμα ε, να ε, αναβάλουμε την ψηφοφορία πρέπει να αποφασίσουμε. Και εξάλλου αρμοδιότητα των ε, πολιτικών ομάδων να μεριμνήσουν τόσο ώστε να γνωρίσουν όλες τις συμβαστικές λύσεις και να κάνουν και την πρόταση τους για τη γραμμή που θα ακολουθηθεί στην ψηφοφορία. Θα ακούσουμε μια τελευταία παρέμβαση από τον κύριο Μπρόκ. Πότε θα πάρει απόφαση η ΙΝΤΕ. That is the only decisive... Αυτό είναι που θα ε, έχει ε, καταληκτική σημασία. Αν τελικά είναι υπερβολικά, ε, αν έχουμε αργήσει υπερβολικά ή όχι. Δηλαδή, ρωτάω πότε ε, έχει προβλεφθεί απόφαση στην ΙΝΤΑ για να ξέρουμε αν μπορεί να αναβληθεί η ψηφοφορία. Μάιο. Συγγνώμη, πριν τις 7 ε, Μαΐου δεν έχουμε εμείς ε, συνεδρίαση. Απάντηση. Δεν είμαι σίγουρη, αλλά έχω την εντύπωση ότι πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει εμείς μέχρι τη 15 Απριλίου. Τότε αναμένεται να ε, διαβάσουμε τη γνωμοδότησή μας στην Ίντα δεν είμαστε η ε, αρμόδια επιτροπή και δεν μπορούμε να το αποφασίσουμε εμείς, κύριος Μπροκ. 15 Απριλίου είναι η προθεσμία για τις τροπολογίες για τα μέλη της ΙΝΤΑ. Πολύ σύντομο το διάστημα. Δεν νομίζω να σας κατάλαβα. Ε, σας είπα ότι 6 και 7 Μαΐου ψηφίζει η ΙΝΤΑ. Ναι, εμείς πότε συνεδριάζουμε και πάλι. Εννοείται για την Επιτροπή Απασχόλησης. Γιατί δεν ψηφίζουμε στις 16. Είναι τρεις εβδομάδες πριν από την ίντα. Μα δεν μπορούμε να αλλάξουμε την ημερομηνία που μας έδωσε η ίντα. Πρέπει να τηρήσουμε την προθεσμία γιατί θα δημιουργηθεί χάος. Και μία μέρα θα έφτανε. Ε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Στο, κυρία Στάινου. Κυρία Πρόεδρε, έχουμε τη σημερινή ημέρα ψηφοφοριών. Την επιλέξαμε μεταξύ των συντονιστών. Και τώρα, μόνο επειδή υπάρχουν κάποιε εσωτερικέ επικοινωνιακέ δυσκολίε σε μια πολιτική ομάδα, να πάμε να αλλάξουμε το χρονοδιάγραμμα, δεν συμφωνώ. Εμείς, η δική μου πολιτική ομάδα, ήταν εις θέση μια χαρά να συζητήσει και τα τελικά αποτελέσματα της προσπάθειας. Και οι πλέον έμπειροι συνάδελφοι γνωρίζουν ότι συχνά είναι αναγκαίο να γίνουν προσπάθειες συμβασμού μέχρι και την τελευταία στιγμή και το τελευταίο λεπτό. Αυτό συμβαίνει συχνά. Και γίνονται διαπραγματεύσεις και για λεπτομέρειες ώστε να επιτύχουμε την μέγιστη δυνατή ε, συνένεση και πλειοψηφία. Γι' αυτό επιμένουμε να γίνει η ψηφοφορία τώρα. Καλώς, θα αρχίσουμε τότε. με το συνδέεται ο κύριος Μάριον Χάρκιν. Τροπολογία 107 ε, ε αποσύρεται και θα αρχίσουμε με την τροπολογία 6. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Ε, ε, ηλεκτρονικός έλεγχος παρακαλώ. Ψηφίστε. Πέρας. Κυρία Σαρτιέ, έχετε πρόβλημα με την κάρτα σας. Ε? Επειδή υπάρχει μόνο μία ψήφος διαφορά, θα επαναληφθεί η ψηφοφορία. Αρχίζουμε και πάλι από την αρχή. Τροπολογία 6. Ψηφίστε παρακαλώ. Δύο υπεράριθμοι ΕΛΚ και δύο υπεράριθμοι στους σοσιαλιστές. Απορρίφθηκε με μία ψήφο διαφορά. Τροπολογία 7 είπε κατά αποχές ε, απορρίπτεται έλεγχος. Πέρας. Περισσεύει ένας από το ΕΛΚ. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 13 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική α υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Πάμε στη συμβαστική Β. Απευθείας. Όχι, όχι, όχι, συγγνώμη, συγγνώμη. Ε, τροπολογία 24 υπέρ. Κατά. Έλεγχος παρακαλώ. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Στο ΕΛΚ πάλι περισσεύει κάποιος. Τώρα. Απορρίπτεται. 25 κατά αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος για την ε, τροπολογία αυτή, παρακαλώ. Ε, για την τροπολογία 25 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίθηκε. Συμβαστική Β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 28 υπέρ κατά Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 28. Ψηφίζουμε. Περάς. Περισσεύει ένας από το ΕΛΚ. Ξέρετε ποιος είναι ονόματα δεν λέμε. 29, ε, όχι, όχι, καταπίπτει. Συμβαστική C. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ε, συμβαστική C. Πέρας. 32 ψήφοι υπέρ. Εγκρίνεται και τώρα. Τροπολογία 43. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 44. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Αρχίζει η ψηφοφορία. και πέρας. Εγκρίθηκε με μία ψήφο διαφορά. Σε 45 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική D υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική ε θέλετε να ελέγξουμε την 55 ε, Πέρας. Δεν απορρίπτεται. Συμβαστική ε υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τώρα 68 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος, μάλιστα. Για την 68. Πέρασε. Περισσεύει ένας από το ΕΛΚ. Αν έχει σημασία, ε, Η 69 καταπίπτει. Συμβαστική F, υπέρ. Αποχές, εγκρίνεται. Η 79 υπέρ κατά αποχές πρέπει να κάνουμε έναν ηλεκτρονικό έλεγχο αρχίζει η ψηφοφορία και εγκρίνεται 81 υπέρ κατά <coughs> αποχές απορρίπτεται Έλεγχος για την 81. Πέρας. Απορρίπτεται 82. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ε, η τερπολογία 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε έλεγχος για την 80 αρχίζει η ψηφοφορία περισσεύει κάποιος από το ΕΛΚ Οκ. πέρασε εγκρίθηκε συμβαστική G υπέρ κατά Αποχές. γκρίθηκε Τροπολογία 96 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Καλώς. Ελέγχουμε την 86. Άρχεται ψηφοφορία. Και πέρας απορρίπτεται 97 όχι καταπίπτει αυτή 98 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 99 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται έλεγχος για την 99 Πέρας. Απορρίπτεται. Η συμβαστική H. Υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Η ε, 105 υπέρ. Κατά. Αποχέ απορρίπτεται. Συμβαστική I. Σας είπα στην αρχή ότι αποσύρεται η 107, οπότε πάμε συμβαστική I, Πέρα. Κάτω. Αποχές εγκρίνεται. Θέλετε έλεγχο για τη συμβαστική ΑΕ. Ωραία. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίθηκε. Εκατόν υπέρ. Κατά. Αστυχές. Απορρίπτεται. 123 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 124 και 125 μαζί υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται Εντάξει, έλεγχος για τις 124 και 125 ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Απορρίπτονται. Ναι. Συμβαστική J. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική K. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 141. σαράντα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος για την 141. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίθηκε. 142 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 143 υπέρ κατά αποχές απορρίφεται 144 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 146 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 145 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 147 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος για την 147 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε με μία ψήφο διαφορά. 148 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 150 Είπε. κατά αποχές έλεγχος Με κρίθηκε. 151 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 156 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 152 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 153 υπέρ κατά αποχές πρέπει να ελέγξουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 154 υπέ Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Πέρας. Απορρίπτεται. 157 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 155 υπέρ. Κατά. Καταπίπτει, συγγνώμη. 155 καταπίπτει. 158 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η πρώτη τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η δεύτερη καταπίπτει τρία, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τέσσερα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται πέντε υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ναι κύριε Μπρόκ θα ήθελα να σας ερωτήσω κάτι νομίζω ξεχάσαμε στην τροπολογία F συμβιβαστική F. Δηλαδή άμεσα κάποια στιγμή ώστε να υπάρξει εγγύηση για το δικαίωμα των κρατών μελών για να νομοθετήσουν. Δεν θα πρέπει να λέει για το δικαίωμα κρατών μελών και Ευρωπαϊκή Ένωση να νομοθετήσουν γιατί σε ε, κάποια θέματα έχει αρμοδιότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει και αυτό να λυθεί υπόψη. Οπότε τι γίνεται εδώ πέρα, με αυτό το λάθος εξαιρούμε ε, αυτούς από τη ρύθμιση. to take immediate steps to guarantee the Άμεσα να λάβει το ώστε να παράσχει εγγύηση για το δικαίωμα των κρατομελών και τη Ευρωπαϊκή Ένωση να νομοθετούν. Τι λέτε, δεν είναι λογικό. Να δώσουμε το λόγο στην κυρία που είναι η συγκεκριά μα τότε, λέει η πρόεδρο. Σα ευχαριστώ. Μιλούμε τώρα για παράθεση του άρθρου 14 της συνθήκης και λέει για το δικαίωμα των μελών να νομοθετήσουν για κάποια θέματα, κρατικές υπηρεσίες, καθολικές υπηρεσίες κλπ. Δεν εξαιρούμε κάποιον, δεν αφήνουμε κανέναν απ' έξω. Απλώς εδώ παραθέτουμε επιλέξει ένα τμήμα, ένα χωρίο του άρθρου 14 της συνθήκης. Ναι, αλλά μιλούμε για κοινωνική νομοθεσία για κάποιες αρμοδιότητες για ποια θέματα ας πούμε για την διάθεση των ε, αποβλήτων αυτό ε, αποτελεί αρμοδιότητα νομοθετική της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλά, ό,τι θέλετε λέει ο κύριος Μπρόκ εκτός είναι προφορική τροπολογία επομένως αυτό το οποίο κάνουμε τώρα μετά την ε, ε, μετά το τι έγινε η ψηφοφορία και πρόκειται επίση για θέμα τη ΣΥΝΤΑ επομένως είναι θέμα τη ΣΥΝΤΑ άρα σας προτείνω να ψηφίσουμε καλά θα ψηφίσουμε τώρα όσον αφορά το σχέδιο γνωμοδότηση όπως τροποποιήθηκε λέει πρόεδρος και τώρα ψηφίζουμε ψήφισε ένας παραπάνω από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα καλώς τώρα και εγκρίνεται με 30 ψήφους υπέρ και 18 κατά. Ανόητη, λέει ο κύριος Μπρόκ. Ε, Τόσο ανόητη. Eh, eh, Στα γερμανικά τρακτός μικρό. Έχω μια ερώτηση προς τον κύριο Μπρόκ, λέει πρόεδρος. Κύριε Μπρόκ. Κύριε Μπρόκ. Σας ρωτώ, θέλετε να μπει στα πρακτικά αυτό το οποίο είπατε πριν. Α, δεν θέλετε. Σας ακούσαμε όμως. Σας... Καλά, όχι. Δεν ακούσαμε τίποτα. Δεν ακούσαμε τίποτα. Καλώς. Συνεχίζουμε την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ευχαριστώ. One is uh, Το επόμενο αφορά τους ναυτικούς. Mm-hmm. E the in mm-hmm. Oh, yeah. Oh, Είστε τώρα έτοιμοι για το σχέδιο εκθέσεως για την πρόταση οδηγίας Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για τους ναυτικούς για τροποποίηση οδηγιών και ακολουθούν οι αριθμοί των οδηγιών. Θα αρχίσουμε με την τροπολογία 39 αυτή έχει αποσυρθεί. Πηγαίνουμε αμέσω στην συμβαστική J. Ψήφι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ακολουθεί παριθμόν 10 και 42 γιατί είναι ταυτόσιμες ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 11 και 43 ταυτόσιμες και αυτές υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται ακολουθούν 12 και 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται Υπάρχουν 13 και 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται και αυτές. Τροπολογία 14 και 46 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Συμβαστική κάπα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 5, τροπολογίες 16 και 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται άρθρο 8 τροπολογία 17 και 51 υπέρ ε, και 18 της αλίας ε, πες 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται συμβιβαστική α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Η 2 της Επιτροπής Αντιείας, ΠΕΣ 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική Β υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η παριθμόν 21 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. ΠΕΣ 5 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται και αυτή συμβαστική C γάμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται θέλετε επαλήθευση λοιπόν ωραία αρχίζει η ψηφοφορία Τέλος. Και όντως απορρίπτεται λόγω ψηφίας. Συγγνώμη, είχε κλείσει η ψηφοφορία και βλέπετε το αποτέλεσμα. Σχόλια χωρίς μικρόφωνο δεν μπορούμε να ακούσουμε. Α, θα επαναλάβουμε τότε γιατί ήταν το μηχάνημα. Πες 7 λοιπόν. Αρχίζει η ψηφοφορία και πάλι. Πες 7. Μία παραπάνω όμως για το σοσιαλδημοκράτες, ε. Ορίστε λοιπόν το αποτέλεσμα. Δεν φταίει η μηχανή. Δεν φταίει η μηχανή λοιπόν. Απορρίπτεται και πάλι. Πες 8. Πες 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική D, δέλτα, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Πέσε νέα αυτή εκπίπτει, τροπολογία 25 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ε υπέρ, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική F, F δηλαδή υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ακολουθεί υπαριθμών 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αυτή υπαριθμών 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται βέβαια κανονικά ψηφίζεται μαζί με την 34 γιατί είναι ταυτόσιμες, άρα και αυτή έχει εγκριθεί. ΠΕΣ 12 δεν ψηφίζεται, συμβαστική G υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. ...36 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική age υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική Ι, αε, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή. Και προχωρώ αμέσως στην τελική ψηφοφορία, διότι δεν ψηφίζεται η αιτιολογική 12. Ψηφίζουμε λοιπόν επί του σχεδίου έκθεσης με ονομαστική ψηφοφορία που αρχίζει τώρα. Ψηφίσατε. Τέλος. 47 ψήφοι υπέρ, 5 κατά και καμιά αποχή. Και τώρα έρχεται η απόφαση μάλιστα για να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις και για το νομοθετικό περιεχομένου ψηφίσματος. Υπέρ, α, νο, όχι, η πρόεδρος λέει ονομαστική ψηφοφορία, αρχίζει η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Αποφασίζουμε τώρα για την ε, απόφαση ψηφίζουμε μάλλον τώρα την απόφαση ε, να αρχίσουν διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 73. ηλεκτρονική πάλι ψηφοφορία αρχίζει τέλος έχετε όλα, όλες τις ψήφους που σας είναι αναγκαίες 51 μάλιστα συνολικά. Yes, please, Κυρία Σαρτιέ, ε, Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τους ε, ε, σκιώδεις όλων των πολιτικών ομάδων. Νομίζω ότι πρόκειται για μια κοινή μας επιτυχία. now vote on the draft opinion Τώρα θα ψηφίσουμε τη σχέδια γνωμοδότησης όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στατικών Επενδύσεων που τροποποιεί μια σειρά κανονισμών. Έχουμε δύο τροπολογίες οι οποίες απεσχέθησαν σήμερα το πρωί. Μιλούμε για την 238 και την υπαριθμόν 284 λέει ο Πρόεδρος. Οπότε και τώρα θα ξεκινήσουμε με την υπαριθμόν 204. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Θα πρέπει να κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίζουμε. Πέρας. Ψηφοφορία. Συμβαστική J. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Διακόσια δέκα πέντε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 216 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 217 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 218 καταπίπτει και προχωρούμε στην 219 ποι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 220 υπέρ κατά αποχές θα γίνει παλιεύση ηλεκτρονική για το 220 ψηφίζουμε πέρας υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 222. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική κάπα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική λάμδα. ελ, Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 230 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 231 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 14 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση ηλεκτρονικά 14. Ψηφίζουμε. Πέρασε Εγκρίνεται. 232. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική. Μ. Μη. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και πάμε κατευθείαν στο 245 λέει πρόεδρος γιατί το 238 κατέπεσε ή επεσήρθη όπως είπαμε στην αρχή ναι επεσήρθη, επεσήρθη 245 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 246 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 247 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 248 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 249 υπέρ, κατά, Απορρίπτεται. 251 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 253 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 250 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 252 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 255 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 254 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 256 υπέρ κατά επαλήθευση Ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε. Ψήφιζε ένας παραπάνω από το ΕΛΚ. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική μη α. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική νη υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και πάμε κατευθείαν στο 269. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 270. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται υπέρ κατά απορρίπτεται 272 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 273 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση ηλεκτρονικά ψηφίζουμε Εγκρίνεται. Συμβαστική όμικρον. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 283. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 282. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 284 έχει αποσυρθεί, οπότε πηγαίνουμε στη συμβαστική π. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 289. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε. Πέρας. Και εγκρίνεται. ένα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 292. Υπέρ. Κατά. Επαλήθευση ηλεκτρονικά. Για το 292. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική Q. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 299 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 300 έλεγχος για το 299 πέρα ψηφορίας απορρίπτεται τοπολογία 300 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται επαλήθευση ηλεκτρονικά ψηφίζουμε πέρας και απορρίπτεται 301 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 302 υπέρ Από κοινού 302 και 306. 302 και 306 υπέρ κατά. Απορρίπτονται. 303 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 304 υπέρ κατά απογές απορρίπτεται 305 υπέρ κατά απογές απορρίπτεται 307 υπέρ κατά αποχέ, απορρίπτεται 308 πρέπει να την ψηφίσουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 309 καταπίπτει. Όχι, πρέπει να την ψηφίσουμε. Υπέρ της 309 κατά απορρίπτεται 310 υπέρ α συγγνώμη γιατί πρέπει να καταπέσει και πάμε στο 312 λοιπόν πρέπει να ψηφίσουμε υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 313 υπέρ κατά Τα 316 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 315 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 14 υπέρ κατά εγκρίνεται 317 υπέρ κατά απορρίπτεται 318 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 319 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 320 υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση του 320. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική ρο. Άρα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 325. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 326. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση ηλεκτρονικά. Για το 326. Υπέρ. Α, συγγνώμη, πέρα στις Δεν κρίνεται. 328. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική σίγμα α, SA υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. Α, συγγνώμη λέει πρόεδρος. Ας κάνουμε την επαλήθευση. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Πέρασε ο Α, όχι, μάλλον, μάλλον ήταν ευρεία η πλειοψηφία, αλλά ορισμένοι δεν έλαβε μέρος στην ψηφοφορία. Άρα πάμε στη συμβαστική S. Σίγουρα υπέρ κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 334 υπέρ κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 336 υπέρ κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 338 υπέρ κατά απορρίπτεται 341 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 342 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται για το 342. Παλήθευση, πέρας και απορρίπτωται Το 343 υπέρ, κατά, αποχές, το 344 υπέρ. Κατά. Η επαλήθευση είναι για το 344. Εγκρίνεται. 345 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 346 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 347 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 348 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 349 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 350 υπέρ κατά αποχές απορρίπτωση 351 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται επαλήθευση για το 351 Ψηφίζουμε. Έχετε ψηφίσει όλοι. Για το 351. Επαλήθευση ηλεκτρονικά. Πέρα ψηφοφορίας. Και εγκρίνεται η τροπολογία 352. Υπέρ. Κατά. Αποχές απολύτω. 353. Υπέρ. Κατά. Αποχές απολύτω. 354 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 354 πέρας εγκρίνεται με ευρία πλειοψηφία 355 καταπίπτει και πάμε στο 356 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 357 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 358 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται για 358 επαλήθευση ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε. πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 359. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 360. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 361 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 362 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται επαλήθευση για το 362 Πέρα της εφορίας. Απορρίπτεται. 363 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 364 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 365 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 266 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 267 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική α. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται υπαλλεύση για το 27 υπέρ ψηφίζουμε και πέρας α 28 υπέρ κατά Άποχες. Απορρίπτεται. 29. Υπέρ. Κατά. Θα πρέπει από αυτού να γίνει επαλήθευση. Το 29. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική β. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Περισμόν 2 στη σελίδα 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Επαλήθευση για το 39. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική BA, β' υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική C, γ, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται πενήντα ένα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 52. δύο υπέρ Κατά. Για να ξανακάνουμε την 52. Πρώτα έκλεισε και η φωνή μου. 52. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 53. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 54 τώρα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και αυτή. 56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 58 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 59 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται α, επαλήθευση επαλήθευση για την 59 αρχίζει η ψηφοφορία ηλεκτρονικά Τέλος. Εγκρίνεται λοιπόν. Τροπολογία 60. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ας κάνουμε όμως ηλεκτρονική επαλήθευση. Αρχίζει τώρα. Τέλος και απορρίπτεται όντω. Η παριθμόν 61 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 62 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 65 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 63 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ακολουθεί η συμβαστική δέλτα D υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ναι, ναι. Λοιπόν. Πρέπει να σηκώνετε καλά τα χέρια. Υπάρχει βέβαια ακόμα πολλή δουλειά να γίνει. Συμβαστική ε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 91 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 92 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 93 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 96 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 94 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 95 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 97 υπέρ κατά αποχές καλύτερα να επαληθεύσουμε με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Αρχίζει. Τέλος. Απορρίπτεται. 98 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 99 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται υπαριθμών 100 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 101 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται υπαριθμών 112 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 113 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Α, επαλήθευση για την 113 αρχίζει τέλος και έχει απορριφθεί 114 υπέρ κατά αποχής εγκρίνεται επαλήθευση καλά 114 λοιπόν αρχίζει η ψηφοφορία τέλος απορρίπτεται Έτσι και αλλιώς κερδίσατε. 116 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται υπαριθμόν 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 117 υπέρ α όχι αυτή εκπίπτει εκπίπτει 117 115 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται στη σελίδα 29 τώρα τροπολογία 136 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 135 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται επαλήθευση επαλήθευση 135 αρχίζει η ψηφοφορία τέλος εγκρίνεται τροπολογία 7 Α, αυτή εκπίπτει. Μάλλον όλες μέχρι την 137. Ψήφι λοιπόν υπέρ της 137. Κατά, αποχές. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει ηλεκτρονική επαλήθευση. Αρχίζει η ψηφοφορία. Εκατόν τριάντα Τέλος και εγκρίθηκε. Ακολουθεί 138 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 139 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Επαλήθευση. Καλά λοιπόν, 139 επαλήθευση. Τέλος. Απορρίφθηκε. 140 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τσεκ. 140. Αρχίζει η ψηφοφορία, 140. Τώρα κλείνει και εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή. Συμβαστική age υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική age A ή τα α δηλαδή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 151 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται θέλετε επαλήθευση λοιπόν 151 αρχίζει η ψηφοφορία τέλος εγκρίνεται Τροπολογία 152 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 155 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 153 Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 154 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 160 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 158 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 156 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται επαλήθευση επαλήθευση για την 156 αρχίζει η ψηφοφορία τέλος και εγκρίνεται 157 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 159 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 161 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Α, επαλήθευση για την 161. Αρχίζει η ψηφοφορία. Τέλος. Πρόκειται για ισοψηφία, άρα απορρίπτεται. Υπαρχούν 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 162 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 164 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 163 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 165 υπέρ Α, όχι, αυτή εκπίπτει. Άρα προχωρώ στην 166 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 167 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 168 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Επαλήθευση. 168. Αρχίζει η ψήφος. Τέλος. Και όντως απορρίπτεται. 169. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 170. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 173 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται επαλήθευση καλά λοιπόν 173 ηλεκτρονική επαλήθευση αρχίζει τέλος οπ λέει η πρόεδρος πραγματικά εγκρίνεται 172 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται επαλήθευση 172 αρχίζει η ψηφοφορία τώρα τελειώνει και εγκρίνεται. 174 υπέρ. Α, όχι, όχι, αυτή εκπίπτει. Άρα, συμβαστική Ι, I, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ακολουθεί υπαριθμόν 182 στη σελίδα πια 34 του κειμένου και έχετε άλλες, άλλη αριθμίση σελίδων οι διάφορες πολιτικές ομάδες. Λοιπόν, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 183. 4 και 5 όλες αυτές μαζί ωραία λοιπόν μαζί υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 186 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 190 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή με συγχωρείτε, εννοώ απορρίπτεται λέει πρόεδρος. 187 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 188 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 189 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 191 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αυτή 193 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 192 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 194 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 195 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 198 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 196 αυτή εκπίπτει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 με ηλεκτρονική ψηφοφορία που αρχίζει τώρα και τελειώνει 35 ψήφοι υπέρ 6 κατά Α, δεν μπορέσατε να ψηφίσετε κυρία μου Να επαναλάβουμε την ψηφοφορία Καλά λοιπόν Ψηφίσατε. Να κλείσουμε τότε την ψηφοφορία. 37 ψήφοι υπέρ, 6 κατά και οι αποχές. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις πολιτικές ομάδες που συνεργάστηκαν σε αυτή την επιταχυμένη διαδικασία. Ζητούσαμε διαρκώς ε, τη συμβολή τους. Σας ευχαριστώ όλους, ευχαριστώ τους και όλους τους ε, και τους συμβούλους go to the draft uh, Τώρα περνάμε στο σχέδιο γνωμοδότησης σε σχέση με το Φόρουμ Οικονομικής Διακυβέρνησης, Απολογισμός και Προκλήσεις, συμβαστική F, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 4, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται συμβαστική β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 23 Καλώς, ε, συμβαστική δέλτα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε τροπολογία 20 τροπολογία 23 διορθώνει ο πρόεδρος τροπολογία 26 Μάλιστα, τώρα ξέρουμε. Πρέπει να ψηφίσουμε για την τροπολογία 24. Για το υπόλοιπο κομμάτι. Ε, τροπολογία 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έλεγχος για την τροπολογία 24. Τέρας. Περισσεύει κάποιος από τους σοσιαλιστές. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 26 είπε κατά Αποχές. Εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 27. Όχι. Συμβαστική C. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 41. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική R υπέρ Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 46. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική ε υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 60. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 61. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα πρέπει να γίνει μια επαλήθευση. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Απορρίπτεται. Ακολουθεί 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβαστική G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική H υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 76 είπε, κατά αποχές απορρίπτεται. Η 77 είπε, κατά αποχές απορρίπτεται. 78 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 79 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε έλεγχος πέρας εγκρίθηκε Συμβαστική J. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική I. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική K. Υπέρ. Αποχές εγκρίνεται. 92 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 93 94 μάλλον υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική M υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Συγγνώμη. Όχι, δεν απε, εγκρίθηκε. Τροπολογία 96, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική L, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 108. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 108 ήταν. Βεβαίω. Να κάνουμε μια επαλήθευση για την 108. Ψήφιστε παρακαλώ. Πέρας. υπέρ. Ναι, ναι. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 120 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 121 υπέρ. Ε, 121 και 122 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 133 και 134 μαζί. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Συμβαστική αν υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Η συμβαστική Q υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Συμβαστική O. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική Π. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 139 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Επαλήθευση για την 139. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 140 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Οκ. Okay, ελεγχός για την 140. Αρχίζει η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται συμβαστική S υπέρ κατά Αποχέ συγκρίνεται. συμβαστική A υπέρ κατά Αποχή συγκρίνεται. τελική ψηφοφορία για το σχέδιο της όπως τροποποιήθηκε. Ονομαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία, παρακαλώ ψηφίστε. Πέρας. πρόβλημα υπάρχει. κυρία Μωρά Σατιέ, ε, άκουσα στη γαλλική μετάφραση με ανάταση χειρός ότι θα ψηφίζαμε. Μπορεί να, ε, αυτό να παραπλάνει σε κάποιους συναδέλφους. Είναι ονομαστική ψηφοφορία. Παρακαλώ να επαναληφθεί. Μάλιστα, λέει ο Πρόεδρος. Τελική ψηφοφορία ονομαστική για αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά, παρακαλώ. Ψήφισαν όλοι. Ωραία, πέρασε. Ωραία. Εγκρίθηκε με ισχυρή πλειοψηφία. Ευχαριστώ. Yes, are you ready? Είστε έτοιμοι για την επόμενη ψηφοφορία? Are you all ready for the vote? σε για την ε, ψηφοφορία για το σχέδιο γνωμοδότησης ε, για ε, τον προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό. Λάουρα Αγγέα, 176 τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 177 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται.

Έλεγχος. 178. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 179. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. <coughs> 180 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 181 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παρακαλώ. Την ελέγξαμε την 181. Α, συγγνώμη, ελέγχουμε την 181. Υπέρ. Ε, ψηφίστε. Πέρας. Και εγκρίθηκε. 182. Υπέρ. Κατά. Αποχές. <coughs> Απορρίπτεται. Έλεγχος. Ψηφίζουμε. Πέρας. Όντως απορρίπτεται. Η 183 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν σηκώνετε τα χέρια. Πρέπει να ξαναρχίσουμε από την αρχή. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 184 υπέρ. Α, είναι ταυτόσιμες. Με την 185. Ωραία. 184 και 185 λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Η συμβαστική M υπέρ κατά αποχές συγκρίνεται, 16 υπέρ κατά απόχέ απορρίπτεται έλεγχος για τη 16 Άρα ε, αρχίζει η ψηφοφορία πέρας εγκρίθηκε συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική ο, ο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε Ανθρωπολογία 20 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 189 και 23 μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 190 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έλεγχος για την 190. Πέρας. Εγκρίνεται. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική π υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ε, συμβαστική Q υπέρ. Κατά Αποχές. Απορρίπτεται. Όχι. Όχι. Συγγνώμη. Εγκρίνεται. Το αντίθετο είναι. 192. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Σημαντική R. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα συμβαστική S υπέρ κατά Αποχέ. εγκρίνεται συμβαστική T υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 29 και 199 είναι ταυτόσιμες, τις ψηφίζουμε μαζί υπέρ. Κατά αποχές πρέπει να γίνει επαλήθευση. Ψηφίζουμε για αυτές τις δύο. 29 και 199 αυτές ψηφοφορίες Απορρίπτονται. 20 πέρα κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 31 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ε, 32 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Συμβαστική U. Α, όχι, έλεγχος για την 32. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται, ναι. Συμβαστική U, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική V υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Σημαντική W υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Σημαντική X υπέρ κατά Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 38 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Είτε τροπολογία 39 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος για τη 39. Πέρας. Ναι, εγκρίθηκε. Ε, συμβαστική Y. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δύο έντεκα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές Συμβαστική Z υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτε 44 υπέρ κατά αποχές 2.13 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική ε, διπλά αλφα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 2.16 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική αλφαβήτα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 47 και 2 19 υπέρ. Α, και η 220. Όχι, μόνο η Σαρδελφάκη 219 υπέρ. Κατά. αφοχές απορρίπτονται. Η 220 μόνη της υπέρ. Κατά. αφοχές απορρίπτονται. Συμβαστική A6 Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική AD. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική AE. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2. 25. Υπέρ κατά α είναι ταυτόσιμη με την 226 μαζί θα τις ψηφίσουμε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τώρα πάμε στην τροπολογία υπαριθμών 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 51 υπέρ κατά απορρίπτεται. Συμβαστική α θ. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 53. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 54. Και μαζί 228. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 229 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 230 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 230 επαλήθευση. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 56. 56, 232 και 231 από κοινού. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 233 υπέρ. Κατά. Α, αποχές. Εγκρίνεται. 234 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 57 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 57. Επαλήθευση. Πέρας. 58 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική AG. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Those in favor, those against. AH υπέρ κατά αποχές και εγκρίνεται. 60, those in favor. 60 υπέρ. Αποχές απορρίπτεται. 61 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 38 έχει υποσχεθεί και πάμε στο 62 ή υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβεστική α, ι, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Εξήντα τέσσερα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 240 υπέρ Κατά. Απορρίπτεται. 65 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 66. Πρέπει να το ψηφίσουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 67. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 68 υπέρ αποχές απορρίπτεται 68 Εγκρίνεται. 69. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Α, απορρίπτεται. 70. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 241. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Επαλήθευση για το 241. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 71. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 72. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 33 λέει πρώτο, ενώ 73. Υπέρ, κατά, Αποχέ. απορρίπτονται. 73, διορθώνει τώρα. Amendment 242, those in favor, against. 242, υπέρ, κατά, Αποχέ, συγκρίνεται. 74, υπέρ, κατά, Αποχέ. συγκρίνεται. 75 υπέρ κατά και απορρίπτεται 76 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 243 those in favor against abstentions carried ε, εγκρίνεται 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται για το 78 πρέπει να γίνει επαλήθευση ψηφίζουμε πέρας εγκρίνεται Το 240 καταπίπτει και πάμε στο 79 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 80 81 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 82 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 83 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται επαλήθευση για το 83 ψηφίζουμε πέρας εγκρίνεται και συμπαθάτε με λέει πρόεδρος 84 Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ε, amendment 85. Ε, those in 85. Υπέρ. Against. Abstention. Αποχές. Θα πρέπει να γίνει ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορία. Oh, it's carried. Amendment 86, those... Εγκρίνεται το 85 επομένω. Πάμε στο 86 υπέρ. Abstention. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Επαλήθω για το 86. And the vote is now closed. Πέρασε ο φορείος. Εγκρίνεται. 87 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 88 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 89 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 90 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 91 υπέρ κατά αποχε εγκρίνεται 92 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 245 υπέρ κατά αποχε εγκρίνεται 90 3 καταπίπτει 94 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 95 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 96 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 97 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Εντάξει, υπέρ κατά απορρίπτεται εκατό, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 101 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 102 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 103 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 104 υπέρ κατά Απορρίπτεται. 105 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση για το 105. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. 106. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 107 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 108 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. 108 υπέρ. Ψηφίζουμε. Πέρασε ο φορείς και εγκρίνεται 109 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική AJ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 111 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 112 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 113 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 114 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 115 υπέρ κατά Εγκρίνεται 116 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται 117 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 247 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 248 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 118. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 119. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 120. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Για το είναι επαλήθευση. Ποιοι είναι υπέρ. Όχι, πρόκειται περί το 120 διορθώνει. 120. Επαλήθευση. Ε, Πέρα στις προφορίες. Εγκρίνεται. Εδώ 21, υπέρ. Κατά. Αποχέ, Απορρίπτεται. 122 και 123 απορρίπτονται. Ε, αποσύρονται, συγγνώμη. Πάμε στο 124 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 125 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίδε. 126 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 127 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 128 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει εδώ έλεγχος για το 128 ψηφίζουμε πέρας απόρριψη όλα αυτά για το 128 λέει πρόεδρος 249 Amendment 249. Υπέρ. Κατά. Α, αποχές εγκρίνεται 129 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 250 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 251 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 252 υπέρ Κατά αποχές εγκρίνεται. 130 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 131 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 132 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 133 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 134 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 135 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 136 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται υπαριθμόν 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 137 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 138 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση για το 138 Πέρας. Και εγκρίνετε; Συμβαστική α. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 141. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 141 επαλήθευση. Πέρας. Εγκρίνεται. Με μια ψηφό για τώρα. Πάμε στην τροπολογία 142, η οποία καταπίπτει. Και πάμε στην υπαριθμό 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 143 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 144 υπέρ α καταπίπτει α όχι δεν καταπίπτει Δεν 144 πρέπει να ψηφιστεί ποιοι είναι υπέρ του 144 κατά αποχές εγκρίνεται 145 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. βασική Β είπε. κατά αποχές εγκρίνεται. 149 είπε. κατά αποχές απορρίπτεται. Καλά, ας κάνουμε μια επαλήφθηση, δεν ήταν σαφές το αποτέλεσμα, 149. Πέρα. Εγκρίθηκε μια ψήφο διαφορά. 150. Υπέρ. Όχι, καταπίπτει. Καταπίπτει. Συμβαστική C. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαναλαμβάνουμε, δεν σηκώσατε αρκετή τα χέρια υπέρ της συμβαστικής C. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 152 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 153 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική D υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ε υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική F. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 161 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 162. Με μια προφορική τροπολογία Αντικαθιστούμε το 7 με 5 στο κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 163 υπέρ. Κατά. <clears throat> Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική G υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Εκατο... ε, συμβαστική H υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική. Άι. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική J. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 171 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. σημαστική K υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ελιπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 175 τώρα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τώρα θα ψηφίσουμε για το ε, σχέδιο γνωμοδότης όπως τροποποιήθηκε. Αρχίζει η ψηφοφορία. Παρακαλώ. Πέρασε. 49 ψήφοι υπέρ. Νομίζω ότι το κερδίσαμε το, με τον ιδρώτα μας ε, το μεσημεριανό διάλειμμα. Θα, θα ξαναπούμε το μεσημέρι. Πιστεύω ότι θα έρθετε πολύ και θα γίνει μίνι σεμινάριο για την παιδική φτώχεια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για όσους συμμετάσχουν στη συζήτηση αλλά και για τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής. Τα λέμε σε κάνα δύο ωρίτσες. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή στο μαραθώνιο ψηφοφορίας. Κυρία Μωρά Σαρτιέ, ευχαριστούμε Πρόεδρε σε εσά, ε, διότι είναι και δύσκολο να προεδρεύει κανείς ένα τέτοιο μαραθώνιο. Τρεις ώρες ε, ε, μας καθοδηγούσατε για την ψηφοφορία, ήσασταν εξαιρετικοί. Ευχαριστούμε και εμείς.